Καλημέρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε και ας μην είμαστε πολλοί. Φαντάζομαι είστε λίγοι και καλοί. Συνάδελφοι, σύμφωνα με την αναβαθισμένη δυνατότητα να έχουμε περισσότερε εκθέσει πρωτοβουλία. συζητάμε την έκθεση του κύριου Τάραντ. Πλαίσιο ΟΗΕ και Σύμβαση για την Αλλαγή του Κλίματος. σύμβαση πλαίσιο του ΟΗΕ. Αρμόδια καθήλυν είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η δική μας υποεπιτροπή εστιάζεται στο θέμα της ασφαλείας. Κρίσεις που δημιουργούνται από την αλλαγή του κλίματος και φυσικές καταστροφές. αναφέρεται και στην Ευρωπαϊκή Στατηγική Ασφαλείας του Δεκεμβρίου του 2008. Κύριε Τάραντ, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την, το θέμα σας. Πράγματι, μπορούμε να πούμε ότι η αλλαγή του κλίματος αφορά περισσότερο την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εγώ πώς το προσεγγίζω το θέμα. Δεν θα συζητήσουμε κατά πόσο συμβαίνει ή όχι η αλλαγή του κλίματος. Συμβαίνει. Και δεν κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αποφύγει. Οπότε είναι και, η ώρα να γίνει κάτι. Να γίνει κάποιος σχεδιασμός Ίσως και να υπάρχουν κάποια μέτρα ανάγκη που θα σχεδιαστούν για να αντιμετωπίσουμε τα επερχόμενα γεγονότα. Σε αυτή την έκθεση ξεκίνησα από παραδείγματα πασίγνωστα στον κόσμο. Δεν θα αναφερθώ σε πλημμύρες, ε, τυφώνες, εξαφανίσεις παγετώνων και την συνεπαγόμενη αύξηση της στάθμης των ωκεανών αλλά θέλω να δω τι μπορεί να κάνει, τι έχουμε στη διάθεσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη και πώς μπορούμε με τους διαθέσιμους πόρους, αν αρκούν, να κάνουμε κάτι. Πώς να χρησιμοποιηθούν οι πόροι μας σε περιπτώσεις ε, ανθρωπιστικών ε, καταστροφών που ίσως να εξελιχθούν και σε βίες συγκρούσεις λόγω ελλείψος τροφίμων, έλλειψης νερού και ε, συνεπαγωμένων ε, μεταναστευτικών ε, φαινομένων. Πρέπει να απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις στην έκθεση. Θέλω να αφαιρθώ σε μερικές από αυτές. Σε ποιο βαθμό οι υφιστάμενες στατικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τα δόγματα και οι έννοιες αντιμετωπίσεως των κρίσεων σχετικά με τις κρίσεις που δημιουργεί η αλλαγή του κλίματος και τα καταστροφές πώς μπορούν να λειτουργήσουν, σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν όλα αυτά να... Το διακυβερνητικό πάνελ για την αλλαγή του κλίματος και οι αναλύσει που έχουν γίνει να ενταχθούν στη στρατηγική προσέγγιση Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ούτω ώστε να δοθεί κάποια συνέχεια πρακτικής φύσεως και να ληφθούν ιδέε αποφάσεις. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, στατιωτικές δυνατότητες, πολιτικές δυνατότητες, παράλληλη χρήση αυτών, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες ανάγκες από τις κρίσεις που προέρχονται την αλλαγή του κλίματος, σε ποιο βαθμό μπορεί να υπάρχει μακροχρόνιο σχεδιασμός, μεθοδολογίες, ανάπτυξη δυναμικού ε, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα αυτές οι ανάγκες. Τρίτον, σε ποιο βαθμό υπάρχει επαρκής συνεργασία στο Συμβούλιο μεταξύ Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεως σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο πραγματικών δυνατοτήτων. Για την ώρα έκανα κάποιες έρευνες, είδα τι γίνεται σε κάποια, σε κάποια στοιχεία, σε κάποιες συνιστώσεις της ε, περίπλοκης θεσμικής μας αρχιτεκτονικής και είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς σφαιρικά την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ενώσης στο σύνολό της. Που ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το θετικό καθήκον ε, και σκοπός αυτής της ε, εκθέσεως. Τι άλλο ήθελα να πω... Μάλιστα. θα ήθελα να υπογραμμίσω και κάτι. Οι απειλές που δημιουργούνται από την αλλαγή του κλίματος, που είναι πολλαπλασιαστικός παράγων, κρίσεων που ήδη υπάρχουν σε κάποιες περιοχές του κόσμου, Βόρεια, Αφρική, Σαχέλ και σε άλλες περιοχές, αυτές οι απειλές είναι πολύ προβλέψιμες. και εύκολα θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε την αντιμετώπιση τους. Δεν είναι τόσο εύκολο να προβλέψει κανείς ακριβώς πότε οι Βόρειοι και οι Νότιοι Σουδανοί θα πολεμήσουν για πετρελοπηγές. Αλλά όσον αφορά τα αγροκτήματά τους και λοιπά, εκεί είναι πιο εύκολο να προβλέψουμε που θα υπάρξουν προβλήματα και συγκρούσεις. και τη χρήση γεών. Τονίζουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία πολιτικού τομέα και στρατιωτικού τομέα. Όμως, όλος μηχανισμός δεν λειτουργεί σωστά κατά την άποψή μου. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη, κάποια καχυποψία από πλευρά μη κυβερνητικών οργανισμών έναντι εμπλοκή των στατιωτικών. Απ' την άλλη, γνωρίζουν πολύ καλά ότι η κοινωνία των πολιτών η ίδια δεν έχει τεχνολογίες, πόρους, εξοπλισμό, μηχανήματα, αεροσκάφη, αεροπλανοφόρα. Μπορούμε να πάρουμε και άλλο παράδειγμα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε. Μετά το τυφώνα Κάθριν, Κατρίνα, η Νέα Ορλεάνη ανοικοδομήθηκε από μηχανικούς του στρατού, διότι οι η πολιτική, ο πολιτικός τομέας δεν είχε το δυναμικό να το κάνει. Νομίζω ότι χρησιμοποίησα το δεκάλεπτό μου. Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσα να πω. Κλείνοντας όμως, θα έλεγα ότι περιμένω οι συνάδελφοί μου να συμφωνήσουν με μένα. Δηλαδή ότι αυτό το θέμα αφορά ακριβώ τη δική μας υποεπιτροπή και αν όχι εμείς τότε ποιος άλλος θα μπορούσε να ασκήσει κάποιες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους φορείς αρμοδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έπρεπε κανονικά να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν είναι μόνο κάτι σημαντικό, αλλά προβλέπεται και συνθήκη της Λισαβόνας. Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Και περιμένω συνεργασία, έμπνευση των συναδέλφων ενδιαφέρον ο πλευράς των μελών αυτής της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον, στους σκιώδεις εισηγητές και μόνο, γιατί μόνο έτσι κι αλλιώς οι εισηγητές είναι παρόντες εδώ σήμερα. Και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Τάραντ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα <clears throat> και η υποεπιτροπή μας θα πρέπει να επιληθεί αυτού του θέματος. Δυστυχώς, σχεδόν έχουμε ξεχάσει τι έλεγε ο κύριος Σολάνα, ο, προ, ο προηγούμενος ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από πέντε χρόνια. Είπε ότι η κλιματική αλλαγή έγινε μια πρώτου μεγέθους πρόκληση ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει αποσπάσει την προσοχή μας από αυτή τη μεγάλη πρόκληση σε άλλα προβλήματα αλλά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Μπαν Κιμούν, είπε το 2009 στο μέσο της χρηματοπιστωτικής κρίσης ότι η ανθρωπότητα έχει λιγότερα από 10 χρόνια για να αποτρέψει την ανεπίστρεπτη κλιματική αλλαγή. Συγκεκριμένα τώρα μας μένουν άλλα 7 χρόνια και σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές και στρατιωτικές πτυχές της κλιματικής αλλαγής είναι τεράστιες οι πτυχές αυτές. Πιστεύω ότι μια πολιτική ασφάλειας θα πρέπει να συμπεριλάβει την κλιματική αλλαγή και τις πιθανές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο και να εφαρμοστεί με τρόπο που δημιουργεί συνέργειες με άλλες πολιτικές. Οι στατιωτικοί αναλυτές, αναλυτές βλέπουν μεγαλύτερους κινδύνους συγκρούσεων, περισσότερη ακυροφροσύνη, περισσότερη τρομοκρατία. Κάθε μέρα που δεν, βλέπουμε, που δεν βρίσκουμε λύσεις στα θέματα αυτά, η αντιμετώπιση της κρίσης θα γίνει πιο πολυδάπανη. Ή πληρώνεται τώρα λίγα ή πολλά αργότερα. Ανησυχώ για το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής δημόσια συζήτηση για αυτό το σημαντικό θέμα. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα σε πρακτικό επίπεδο. Χρειάζεται ανταλλαγή εμπειριών μέσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κομισιόν και οι κύριοι εταίροι σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι χώρε BRICS, η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, η Βραζιλία, φυσικά όλε αυτέ οι μεγάλε χώρε θα πρέπει να συντονίσουν τι δράσει του για την αντιμετώπιση κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μηχανισμό έγκαιρη προειδοποίηση για τι κρίσει που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τι φυσικέ καταστροφέ και επίσης οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τα θέματα αυτά των φυσικών καταστροφών με παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Θα πρέπει να παροτρύνουμε τις χώρες μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν τις δυνάμεις τους πιο αυτόνομες σε σχέση με τη χρήση ενέργειας. Έχει αλλάξει και ο κλασικός ρόλος ενός στρατού που είναι η προστασία από επιθέσεις και εισβολές. Είναι πολύ πιο διαφοροποιημένος ο ρόλος των στρατών και επομένως οι στρατιωτικές δυνάμεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και πολιτική υποστήριξη σε περιπτώσεις μεγάλων απειλών όπως είναι μαζικές μεταναστάυσεις πληθυσμών. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο λοιπόν στη διάθεσή μας πια και αυτή η έκθεση θα μπορούσε να μας βοηθήσει <clears throat> να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα και <clears throat> και να, ε- να ανεβάσουμε την συνειδητοποίηση του πληθυσμού για τα θέματα αυτά. Κυρία Λόζιν, η οποία είναι επίσης σκιώδης εισηγήτρια. <clears throat> Σας ευχαριστώ. Εγώ έχω μεγάλο ενδιαφέρον για να δω ποια θα είναι η γραμμή που θα έχουμε στην έκθεση αυτή γιατί είναι μια έκθεση που την εκπονεί η ομάδα των Πρασίνων. Θέλω να πω επίση ότι η ομάδα μας λέγεται ε, η ομάδα GUE NGL, είναι και πράσινη σκανδιναβική αριστερά επομένω, επομένω τα θέματα αυτά μας ενδιαφέρουν και μας ιδιαίτερα. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δούμε αν θα μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συνένεση ή θα καταλήξουμε σε διαφορετικές απόψει για το θέμα αυτό γνωρίζω πολύ καλά ότι είμαστε βέβαια στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Μας ενδιαφέρει όμως να έχουμε μια συνολική προσέγγιση και δεν θέλω τώρα να σας ε, κατευθύνω προς άλλες πορείες από αυτή η οποία είναι η φυσιολογική για μια επιτροπή όπως αυτή. Αλλά εγώ προέρχομαι από ένα αριστερό, παραδοσιακά αριστερό χώρο και ίσως δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία θα πούν οι άλλοι συνάδελφοι. Η Επιστημονική Επιτροπή της Γερμανικής Bundestag έχει κάνει μια έκθεση για τα θέματα αυτά από την οποία μπορώ και να σας παραθέσω ορισμένα κομμάτια. Λέει η έκθεση αυτή, η οποία έχει αντιμετωπίσει το θέμα της κλιματικής αλλαγής, τα εξής. Λέει ότι τα βιομηχανικά κράτη θα πρέπει βάσει της αρχής ο υπέτειος θα πρέπει να πληρώνει, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και πρέπει να υπάρξει και η ανάληψη ευθύνης για την εξασφάλιση της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο από τα βιομηχανικά κράτη, η οποία θα πρέπει να γίνει και ορατή μέσα στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, η οποία αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια αντιδραστική και κοντόφθαλμη στρατηγική και μόνο. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης για να αποτρέψουμε τις χειρότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Και υπάρχει μια διεκδίκηση να περάσουμε από την στρατιωτική δαπάνη και ανάπτυξη σε προσπάθειες οι οποίες θα βοηθήσουν σε κοινωνικό επίπεδο. Επομένως, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των κρίσεων, αντιμετωπίζοντας τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα στον κόσμο. Αναφέρεται λοιπόν το θέμα της ε, κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών του, αλλά δεν πρέπει να το δούμε μονάχα μονόπλευρα σαν ένα πρόβλημα απειλών. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ε, οικονομικές συνέπειες του, αλλά να δούμε και τι επιπτώσεις θα έχει και τι ευκαιρίες θα μας δώσει για την διατροφή του πληθυσμού του πλανήτη μας. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να δούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για την κλιματική αλλαγή για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια αηφόρα αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζάνκε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση που παρουσίασε ο κύριο ε, Τάρεντ και να κάνω κι εγώ κάποιε υποδείξει από πλευρά μου. Καταρχά να εκφράσω κάποιε αμφιβολίε. Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον ορίσαμε σωστά τον ίδιο τον τίτλο της έκθεσης. Τι εννοώ. Αναφερόμαστε σε δύο πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο πανομοιότυπα. Καταρχάς πρέπει να δούμε τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και διορθώστε με εδώ αν κάνω λάθος, αλλά έχω την αίσθηση ότι η αλλαγή του κλίματος και οι φυσικέ καταστροφές θα πρέπει να είναι ε, Μεγάλη διάρκεια δεν θα είναι κάτι το οποίο θα συμβεί εν μία νυχτή και μετά έχουμε κάποιες περιπτώσεις όπου έχουμε ένα, ε, μία καταστροφή που συμβαίνει σε μία νύχτα. Ένα εξαιρετικά ε, μεγάλο φυσικό φαινόμενο, μια νυχτη και μετα εχουμε καποιες περιπτωσεις οπου εχουμε μια καταστροφη που συμβαινει σε μια νυχτα ενα εξαιρετικα μεγαλο φυσικο φαινομενο μια μεγαλη καταστροφη ε, η αλλαγή του κλίματος λοιπόν είναι μακροπρόθεσμη, αλλά η φυσική καταστροφή είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και μέσα σε μερικές ώρες. στο Κοινοβούλιο αναφερόμαστε εν γέννη στην συνδρομή που μπορούμε να προσφέρουμε σε περίπτωση κρίσεων. Για παράδειγμα, μετά τα όσα συνέβησαν στην Αϊτή ε, ή τι συνέβη στην Ουγγαρία. Ε, σε τέτοιες περιπτώσεις ε, αναφέρονται κάποια επιχειρήματα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν κάποιες επικρίσεις και η αλήθεια είναι ότι ορισμένες φορές όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε φυσικές καταστροφές, δίνουμε πάρα πολλά χρήματα στα θύματα και προσπαθούμε να ανοικοδομήσουμε ε, το τοπίο μετά από την καταστροφή, αλλά μπορεί ε, να μην είναι χρονικά σωστή η βοήθειά μας. Από την εμπειρία που αποκομίσαμε από την ΑΕΤ, για παράδειγμα, ήταν πολύ πικρά τα αποτελέσματα και αυτό έχει σημασία, διότι ε, ο τρόπος με τον οποίο θα δράσουμε καθορίζει πόσοι, άνθρωποι θα επιβιώσουν και νομίζω ότι είναι θεμελιώδου σημασία αυτό που ανέφερε ο κύριο Στάραντ. Δηλαδή οι δυνατότητες που έχουμε και η δυνατότητα να κινητοποιήσουμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Ορισμένες φορές ε, ανησυχώ ότι δαπανώνται πάρα πολλά χρήματα σε ανθρωπιστική βοήθεια Δίνονται πάρα πολλά χρήματα σε αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Ίσως είμαστε ο μεγαλύτερος χορηγός ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δωρητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν θέλουμε να συντονίσουμε τη δράση μας και να κινητοποιηθούμε αμέσως ε, έχουμε πρόβλημα. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν εδώ στην έκθεση να αναφερθούμε λίγο καλύτερα στα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Διότι όταν συμβαίνει μια φυσική καταστροφή, είτε θα διαθέτουμε κάποια μέσα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι εκ νέου και δεν υπάρχει χρόνος για κάτι τέτοιο. Για να αποφύγουμε λοιπόν πιθανά προβλήματα όταν ε, συζητάμε τα ίδια τα μέσα και τις υποδομές που ε, διαθέτουμε, ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή ε, το εξής ερώτημα. Έχουμε τη δυνατότητα να δράσουμε μόνο επί χάρτου, όπως μας επικρίνουν πολλές φορές αρκετοί, ε, διότι ορισμένες φορές τα χαρτιά φαίνονται όλα πάρα πολύ ωραία, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη όταν υπάρχει καταστροφή. Νομίζω ότι το θέμα αποτελεί πρόκληση, αλλά είναι και ένα υπαρκτό πρόβλημα. Και χαίρομαι που έχουμε αυτή την έκθεση, διότι υποχρεώμεθα να δώσουμε κάποιες απαντήσεις επί του πρακτέου και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, για όλους. Κατά βάση μας ενδιαφέρει όμως το θέμα της ε, ε, συνεργασίας πολιτικής προστασίας. Ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε κάποιους κανόνες προκειμένου οι στρατιωτικές δυνάμεις αλλά και οι πολιτικές δυνάμεις να μπορέσουν να δράσουν και να συνεργαστούν, αλλά κατά την άποψή μου υπάρχει και ένα ακόμα θέμα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη, είναι η πρόληψη σε αυτή την έκθεση. Τώρα, όταν δρούμε κατά τη διαχείριση της κρίσης ε, για το θέμα των φυσικών καταστροφών, νομίζω ότι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε όταν υπάρχει φυσική καταστροφή και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, καταστάσεις που δεν αφορούν μόνο ένα κράτος μέλος, αλλά και πολλά κράτη-μέλη. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να βοηθήσουμε δύο ή τρία κράτη-μέλη. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε και κάτι για να ε, μειωθεί το κόστος της καταστροφής. Διότι αν εξετάσουμε λίγο τα πράγματα πιο προσεκτικά, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν πλημμύρες, υπάρχουν σεισμοί. Έχουμε τυφώνες, ε, όχι στην Ευρώπη, αλλά έχουμε και τη, αντίστοιχα φαινόμενα στην Ασία και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα εξασφάλισης αυτών των ανθρώπων, ασφάλειας, ώστε να είναι λίγο μικρότερο η ζημιά για αυτούς. Ίσως να έχουμε και ένα κώδικα βέλτιστων πρακτικών. Ευτυχώς υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη τα οποία έχουν μακρά πείρα, έχουν λάβει συγκεκριμένα μέτρα και υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα για να αντιμετωπίσουν φυσικές καταστροφές. Επομένως, ένας οδηγός βέλτιστων πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε ίσως να είναι χρήσιμος, ώστε να εκπαιδεύσουμε και αυτούς οι οποίοι δεν είναι τόσο άρτια προετοιμασμένοι ε, σε αντίστοιχα προβλήματα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την έκθεσή σας και ελπίζω η έκθεση αυτή να μην ε, εξεταστεί μόνο από το ιδεολογικό της υπόβαθρο, διότι χρειαζόμαστε και κάποια συγκεκριμένα μέτρα κοινή λογικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Είναι δύσκολο με αυτό το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα σχόλια που έχετε κάνει. Να σας πω ότι καταρχήν για την κυρία Λέζινγκ καμιά φορά τα κράτη-μέλη ακόμα και σε εποχές οικονομικής κρίσης και λιτότητος εξακολουθούν να δαπανούν πολλά στον αμυντικό τους προϋπολογισμό. Και πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι και μια ευκαιρία να προτείνουμε μια διαφορετική χρήση των στρατιωτικών πόρων μας. Να μην είναι μονάχα σε επιφυλακή για κάτι το απρόβλεπτο, αλλά να μπορούν να συμμετέχουν πιο επωφελώς στη σχεδίαση για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέρχονται από φυσικές κρίσεις ή από κλιματικές αλλαγές κτλ. Και υπήρξαν εδώ και κάποια καλά παραδείγματα. Στην περίπτωση των πλημμυρών στη Μοσαμβίκη πριν από κάμια δεκαετία χρόνια και μπορούν εκεί να χρησιμοποιηθούν στρατιωτικοί πόροι και εξοπλισμός σε ανακουφιστικές ενέργειες. Υπήρξαν όμως και διαφορετικά παραδείγματα όπου για λόγω πολύπλοκων προβλημάτων νομικού και οργανωτικού χαρακτήρα οι στρατιωτικές δυνάμεις δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επωφελώς, παραδείγματος χάρη στην ΑΕΤ, όπου πολλά προβλήματα μπορούσαν να θα μπορούσαν να είχαν επιληθεί πολύ πιο εύκολα με το αμερικανικό ναυτικό παρά με την ε, παροχή βοήθειας από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ. Υπήρξαν όμως και κάποια θετικά παραδείγματα. η αποστολή που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της ΚΕΠΑ για το Σαχέλ. Και υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι πράγματι είναι εμπεριστατωμένη αυτή η σχεδίαση για την αντιμετώπιση της κρίσης εκεί. Θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται και στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα θέματα, όπως είπε και η πρόεδρος της ε, συνεργασίας πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων, ήδη είχαμε την έκθεση Μπαρνία για το θέμα αυτό, όπου προσπαθούσαμε κατά πόσο αυτή η έκθεση εξακολουθεί αυτά τα οποία είχε πει ο κ. Μπαρνιέ εξακολουθούν να είναι έγκυρα ή αν χρειάζονται επικαιροποίηση. Το κύριο ερώτημα το οποίο παραμένει είναι πώς θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τις στρατιωτικές προκλήσεις μέσα στον πλήρη κύκλο προκλήσεων λόγω συγκρούσεων. Η προειδοποίηση, η αντιμετώπιση των κρίσεων, η ανοικοδόμηση και η ε, δημιουργία εθνικών δομών. Η συλλογή πληροφοριών, η ανάλυση των πληροφοριών, ο πολιτικός και σχεδιασμός και διαχείριση των κρίσεων, όλα αυτά είναι στοιχεία που μπορούμε να επωφεληθούμε από τις βέλτιστες πρακτικές και μας ενδιαφέρει επίσης να αναπτύξουμε και ικανότητα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε και μια αναθεώρηση της πρότασης Μπαρνιέ για να δούμε αν μας λείπει κάτι και αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης αυτής είναι η πρώτη εξέταση θα γίνει στις 29 Μαΐου. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι μέχρι τις 20 Ιουνίου. Η δεύτερη εξέταση της έκθεσης 28 Ιουνίου και θα εγκριθεί η έκθεση αυτή στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων το Σεπτέμβρη, κάπου το Σεπτέμβρη και τον Νοέμβριο θα έρθει στην Ολομέλεια. Έτσι προβλέπεται. Έχουμε αρκετό χρόνο για να καταρτήσουμε μια καλή έκθεση. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη η εφαρμογή του θέμα της νομοθεσίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό Καλωσορίζουμε τον εισηγητή και συναδέλφο, τον κύριο Κυρίλοφ, και του δίνουμε το λόγο. Η Ευγένη έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει το σχέδιο αυτό της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ενιός Ευρωπαϊκός Ουρανός, όπως γνωρίζουμε, είναι αρκετά φιλόδοξη η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η όλη ιδέα να δημιουργήσουμε ένα αέριο χώρο πραγματικά έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, ένα αέριο χώρο, είναι κάτι αξέπαινο. Εμείς τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου που πετάμε συχνά ε, διαπιστώσαμε κάποιες θετικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια και είναι μία από τις πρωτοβουλίες που κατά την άποψή μου εξακολουθεί να περνά παρατήρητη τη θέμενη αξία όσον αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν το παρατηρούν. Γνωρίζουμε βέβαια ότι πρέπει να αναπτυχθεί. Είμαστε στα πρώτα στάδια και σοβαρές συμφορήσεις στον εναέριο χώρο της Ευρώπης πρέπει να αποφευθούν. Εδώ στην Υποεπιτροπή ασχολούμεθα με τις, ε, τα αποτελέσματα, τις συνέπειες που έχει αυτή η πρωτοβουλία όσον αφορά το στρατιωτικό χώρο. Η στρατιωτική είναι ο μεγαλύτερος χρήστης του εναερίου χώρου στην Ευρώπη. Με σημαντικά, σημαντικό αριθμό αεροσκαφών, μαχητικών και άλλων, Χρειαζόμαστε τη συνεργασία των στρατιωτικών για να πετύχουμε τους τελικούς μας ε, ε, στόχους. Χρειάζεται μια ασφαλής και ευέλικτη συνύπαρξη των επιχειρήσεων του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Παρά το γεγονός ότι ο κανονισμός για τον εναέριο χώρο, τον ενιαίο χώρο δεν ε, αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την εκπαίδευση, επιβεβαιώνουν τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να λάβουμε πλήρως υπόψη τις ανάγκες που σχετίζονται με την πολιτική, την εθνική σε θέματα άμυνας και ασφαλείας και η στατιωτική χρήση από πλευράς κρατών μελών των εναερίου, του εναερίου χώρου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τον ενιαίο εναέριο χώρο. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην νομοδότηση που συζητούμε. Εδώ υπογραμμίζουμε τη σημασία που έχει ο ομαλός συντονισμός θετικού και πολιτικού τομέα και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η σχετική νομοθεσία και η εφαρμογή αυτής ε, θα πετυχαίνει αυτό το στόχο. Λαμβάνοντας υπόψη ε, ποιε είναι οι συνέπειε τη προσπάθεια που καταβάλουμε στο δυτικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλεία πολύ σύντομα, ε, συγγνώμη, πρόσφατα στο ΣΥΖΑΡ ε, εκλήθη να γίνει πιο δραστήρια. Αυτό είναι ο τεχνικό κλάδο και ο κλάδο έρευνα τη πρωτοβουλία. Και αυτή η εντολή θέλει αξιολόγηση συνεπειών του ΣΥΖΑΡ για την αμυντική κοινότητα και θα πρέπει να υπάρξει ένα βήμα όπου θα συμμετέχουν όλοι οι στρατιωτικοί φορείς στις συζητήσεις. Το Eurocontrol, το ΝΑΤΟ ε, συνέβαλαν στο κείμενο που συντάσσω ε, και χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ του πολιτικού και τομέα. Χρειάζεται καλύτερη διαλειτουργικότητα, χρειάζεται κοινή υποδομή. Αποτέλεσμα, θα είναι σημαντική περικοπή των δαπανών, πέρα από τα περιβαλλοντικά ωφέλη. Εκτιμάται ότι η εφαρμογή του ΣΥΖΑΡ στα στρατιωτικά αεροσκάφη και τον έλεγχο εδάφους απαιτεί περίπου 7 δις ευρώ επενδύσεις. Λίγο περισσότερο από 25% του συνολικού ποσού που είναι 30 δις για όλο το πρόγραμμα. Είναι μεγάλη επένδυση κυρίως σε εποχές ε, οικονομικής κρίσεως. Άρα θα πρέπει αυτό να αναλυθεί σε πρώτο στάδιο, σε αρχικό στάδιο, με ρεαλιστικό τρόπο και φευρετικό τρόπο. Χρειάζεται έγκαιρη εφαρμογή του συστήματος. Υπάρχει μια κρίσιμη φάση της αναπτύξεως. Αν δεν δράσουμε συνεκτικά, συντονισμένα, θα είναι μεγαλύτερη απαιτούμενη περίοδος για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος. Και αυτό συνεπάγεται σοβαρές δαπάνες. Η μεγάλη πρόκληση για τους αθλητικούς είναι να επενδύσουν έγκαιρα σε νέες τεχνολογίες, να διαθέσουν χρήματα. Και στη γνωμοδότηση αυτή υπογραμμίζω το ότι πρέπει να βρεθούν γρήγορα τρόποι αντιμετωπίσεως της πρόκλησης για τους στρατιωτικούς, γιατί όπω γνωρίζουμε τα εμπορικά αεροσκάφη ο εμπορικό τομέα ενδιαφέρεται, ο πολιτικό τομέα ενδιαφέρεται και έχει κίνητρα. Κυρίω οι μεγάλε εταιρείε θέλουν να συμμετάσχουν. Οι στατιωτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ε, οικονομικές συνέπειες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, το Eurocontrol, τους διάφορους φορείς που με βοήθησαν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν πολύ καρποφόρα η συνεργασία μαζί μας, ε, και η συζήτηση και ο διάλογος. και με κάνει αυτό να αισθάνομαι αισιόδοξο για την ε, εφαρμογή του όλου προγράμματος, την υλοποίησή του. Και πιστεύω ότι η συνεργασία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων με τους ειδικού του ΝΑΤΟ ε, πήγε αρκετά καλά. Καμιά φορά εμεί οι πολιτικοί περιπλέκουμε τα πράγματα, αλλά μέχρι τώρα η εντύπωσή μου είναι ότι καλά πάμε. Σας ευχαριστώ. μερικές φορές, όχι πάντα. Ευχαριστώ, Ευγένη. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ουμπέρτο Ρώση, το Στρατιωτικό Σύμβουλο μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την υποεπιτροπή που προσκάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητήσουμε αυτό το τόσο περίπλοκο ζήτημα, την εφαρμογή του ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και ιδίως στη σχέση με τη στρατιωτική συνιστόσα για το θέμα αυτό. Θα είναι πρόκληση για μένα να προσπαθήσω να συνοψίσω την παρουσίασή μου για κάτι το οποίο ξεκίνησε το 2000 ε, σε 10 λεπτά. Θα προσπαθήσω όμως και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων εάν ε, ξεπεράσω λίγο το χρονικό περιθώριο που μου δίνεται. Γιατί και πότε ξεκίνησε ο ενιαίος ουρανός. Ξεκίνησε στις αρχές του 2000 διότι τότε ε, αυξάνονταν οι απαιτήσει για τις εναέριες μεταφορές και ε, υποθέσαμε ότι οι υποδομές για να υποστηρίξουν αυτές τις απαιτήσει δεν θα επαρκούσαν για να ανταποκρινθούν στις ανάγκες μας ε, το 2010 και το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ανέλαβε τα ενία και ξεκίνησε αυτή την πρωτοβουλία και τότε η εκδοχή που εξετάζαμε δεν ε, θα μπορούσα να πω ότι ήταν δραματική, αλλά ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, διότι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 27 κράτη-μέλη με διαφορετικά πρότυπα. Ε, το να συντονίσουμε 27 κράτη-μέλη με διαφορετικούς, διαφορετικές προκλήσεις δημιουργούσε φυσικά με μια, μια τεράστια πρόκληση και επομένως ε, ε, υπήρχε και θέμα αποτελεσματικότητας του συστήματος. Πέραν δε αυτού, υπήρχε και ανάγκη να συντονίσουμε, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και από τον κύριο Κυρίλοφ, τους δύο βασικούς παράγοντες ε, στον εναέριο χώρο, το στρατιωτικό και το πολιτικό τομέα, διότι ε, τότε ο εναέριος χώρος που απαιτούνταν από το στρατιωτικό τομέα για τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες ήταν σχεδόν ένα τεράστιο ποσοστό του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου χρησιμοποιόταν με έναν ε, παροχημένο, θέλετε, τρόπο εκμετάλλευση αυτού του εναέριου χώρου, μόνο για στρατιωτικέ ανάγκες. Δεν υπήρχε ουσιαστικά καμία συνεργασία με την πολιτική συνιστόσα τότε. Το πρώτο τμήμα λοιπόν του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού ε, ξεκίνησε τότε, το λεγόμενο CES1, δημιουργήσαμε ένα αρχικό ρυθμιστικό πλαίσιο, αρχίσαμε να εξετάζουμε λίγο τις τεχνολογικές βελτιώσεις ε, που θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε στο σύστημα ε, διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, το ATM, και θέσαμε τα θεμέλια για κάτι το οποίο πλέον ε, είναι εδρεωμένο στην Ευρώπη, ε, ε, την ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου. Πρόκειται για μια πολύ απλή αρχή. Είναι βασικά το γεγονός ότι ο εναέριος χώρος δεν ανήκει ούτε στο στρατιωτικό ούτε στον πολιτικό τομέα, ανήκει στον κάθε χρήστη ανα πάσα στιγμή βάσει των αναγκών του. Το 2004 επιτύχαμε το στόχο μας μεν, αλλά υπήρχε μια αίσθηση ότι το, η αύξηση των μεταφορών και το αίτημα για αύξηση των μεταφορών ήταν τόσο υψηλή που έπρεπε να ε, χρησιμοποιηθούν νέα μέσα. Και επομένως ξεκίνησε η εφαρμογή του CES2, του δεύτερου τμήματος του ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, που βασίστηκε σε πέντε πυλώνες. Ο πρώτος ήταν να εξετάσουμε την απόδοση του συστήματος, ε, του συστήματος διαχείρισης της κίνησης ε, από πλευράς ασφαλείας, περιβάλλοντος, δυνατοτήτων και αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος. Ε, χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν, αναπτύχθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες για την εξέταση αυτών των στοιχείων. Επίσης, ε, βασικό στοιχείο θεωρήθηκε και η τεχνολογία και δημιουργήθηκε το κοινό πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία ΣΕΖΑΡ και υπήρξαν και νέες ε, ε, ε, αρμοδιότητες για την EAS που είναι η υπηρεσία αρμόδια για την ασφα... ασφάλεια. Είχαμε το σύστημα της διαχείρισης εναέρειας κυκλοφορίας στους αερολιμένες. Και τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, εξετάσαμε και τις δυνατότητες που έχουν οι αερολιμένες, διότι το βασικό πρόβλημα συμφόρησης θεωρήθηκαν οι αερολιμένες και όταν έπρεπε να ξεκινήσει αυτή η λεγόμενη αρχή gate to gate. Ένα σημαντικό στοιχείο του 9 ουρανού 2 ήταν ότι θέλαμε να αρχίσουμε να ε, μειώνουμε αυτό τον κατακαιρματισμό που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον ενέωριο χώρο και να δημιουργούμε ξεχωριστά μπλοκ, δηλαδή ομάδες χωρών οι οποίες ε, καθορίζουν κοινού κανόνες με γνώμονα πάντα την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης εναέριων μεταφορών. Δημιουργήθηκε επιπλέον και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο είχε συγκεκριμένες ε, λειτουργίες και θεωρήθηκε ότι το Eurocontrol είναι ο αρμόδιος φορέας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ε, τις ανάγκες ε, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης των Εναέριων Μεταφορών. Να σας πω τώρα και λίγα πράγματα για τη ε, συμμετοχή του στρατού σε όλη αυτή την περίπλοκη συζήτηση. Ο κύριος ε, Κυρίλοφ ήδη αναφέρθηκε στη βασική ανησυχία για τη στρατιωτική πλευρά, ε, όπως την ε, βλέπουμε για τα επόμενα χρόνια. Αυτό αφορά το κόστος για την εφαρμογή της τεχνολογίας ΣΕΖΑΡ για το στρατό. Ο κύριος Κυρίλοφ αναφέρθηκε στο αναμενόμενο κόστος, το οποίο υποτίθεται ότι θα είναι περίπου 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η εκτίμηση έγινε στην αρχική ε, διαδικασία, στο αρχικό στάδιο της ε, διαδικασίας. Πρέπει να σας πω ότι έκτοτε έχουν γίνει αρκετά και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες ε, και στην ΣΕΖΑΡ αλλά και στο Eurocontrol γιατί συνεισέφεραν ιδιαίτερα και μπορέσαμε να διευκρινίσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα ποιες είναι οι επιχειρησιακές ανάγκες αλλά και οι επιπτώσεις ε, ως προς το κόστος για τη συμμετοχή και τη στρατιωτική πτυχές στο ΣΕΖΑΡ. Ε, αυτή την εβδομάδα ο επικεφαλής της Άμενης συναντήθηκε εδώ στο Συμβούλιο με ε, τους αρμοδίους και έγινε μία συζήτηση και βάσει μιας απόφασης που θα πρέπει να εγκρίνουν τα κράτη-μέλη, το κόστος θα μειωθεί σημαντικά. Ε, βεβαίως πρέπει να γίνουν αρκετές συζητήσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ε, εν τέλει, πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία ε, στρατιωτικής και πολιτικής συνιστώσας είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο ευρωπαϊκό ουρανό, ο οποίος θα μπορέσει να καλύψει καταρχάς το αίτημα για κατάλληλες εναερίες μεταφορές για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά να λάβει υπόψη και τα εθνικά αιτήματα, την ανάγκη δηλαδή για ε, επιχειρήσεις ασφάλειας και άμυνας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ε, εξέταση των ε, πτυχών ε, του ενιαίου Ευρωπαϊκού Ρανού 3, CES 3. Και θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία λοιπόν μεταξύ των δύο συνιστοσών θα συνεχίσει να αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της μελλοντική εξέλιξης του προγράμματος. Νομίζω ότι κατάφερα να σας ε, περιγράψω σε πολύ γενικές γραμμές ποια είναι τα βασικά στοιχεία για την ε, στρατιωτική συνιστόσα στον Ενίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω και σε οποιοδήποτε ερώτημά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον σκιώδη συγητή. Σας ευχαριστώ από το ΕΛΚ. Επειδή ο κύριος Κυρίλοφ και εγώ ζούμε σε περιοχές που είναι γεωγραφικά πολύ κοντά μεταξύ τους, πολλές φορές ερχόμαστε μαζί με το αυτοκίνητο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συζητάμε πολύ συχνά. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα σχέδιο έκθεσης το οποίο είναι μεγάλης ποιότητας, υψηλής ποιότητας. Συζητήσαμε επίση και στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση του ΕΛΚ για τα θέματα αυτά και δεν έχουμε καμιά ιδιαίτερη επιφύλαξη για τα ζητήματα αυτά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Κυρίλοφ υπογράμμισε τη σημασία που έχει το να υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση του εναέριου χώρου ώστε και οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικές αρχές, οι συνοριοφύλακες όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια σχέση με το ένα αέριο χώρο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν ενώπιον των πολιτών. Κάτι ακόμα επίσης σε τυπικό επίπεδο. Αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Κυρίλοφ έχει διατυπώσει τη γνωμοδότησή του επί τη βάση του εγγράφου της Κομισιόν και ίσως επί τη βάση μιας μη ε, δημοσιευθήσεις μορφής της έκθεσης της Κομισιόν. Νομίζω ότι μόνο αυτός έχει αυτό το κείμενο της Κομισιόν, το πρώτο, την πρώτη μορφή του εγγράφου της Κομισιόν. Ο εισηγητή τώρα στην Επιτροπή Μεταφορών έχει επίση συντάξει ήδη την έκθεσή του, αλλά δεν είναι ακόμα διαθέσιμη από ό,τι ξέρω. Θα χρειαστούμε επομένω λίγο χρόνο για να έχουμε τη μετάφραση σε όλε τι γλώσσε. και επομένως θα χρειαστεί ίσως να καθυστερήσουμε κατά μία εβδομάδα την ε, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Έτσι θα είναι πιο εύκολο για μας να καταθέσουμε τροπολογίες, αλλά ξέρω... Ξέρω ότι η έκθεση αυτή αντιμετωπίζει και το θέμα της συνεργασίας πολιτικών και στρατιωτικών αρχών για τον ενάριο χώρο Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό, αλλά θα πρέπει να έχουμε τον χρόνο να διαβάσουμε πλήρως την έκθεση και να λάβουμε γνώση όλων των στοιχείων, γιατί θα μπορούσαν να προκύψουν και νέες εξελίξεις στην Επιτροπή Μεταφορών και θα πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν τη γνωμοδότησή μας. Αυτά λοιπόν σε τυπικό επίπεδο θα πρέπει να κάνουμε να καθυστερήσουμε κατά μία εβδομάδα την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Λόιζεν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ βέβαια δεν έχω όλα αυτά τα έγγραφα που αναφέρθηκαν. Το μόνο πράγμα στο οποίο μπορώ να βασιστώ είναι το κείμενο της γνωμοδότησης. Σίγουρα είναι πολύπλοκο το σύστημα αυτό και έχουν παρουσιαστεί οι πάρα, πολλές πτυχές αυτού του συστήματος από τον κύριο Κυρίλοφ. Και επίσης υπάρχει και το σύστημα αυτό το οποίο παρουσίασε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Υπήρχαν στο παρελθόν να χρησιμοποιηθεί και ο χώρος, ο εναέριος που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή από τις στρατιωτικές δυνάμεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι το αναπόδραστο να προχωρήσουμε και σε διαπραγματεύσεις με τις στρατιωτικές αρχές για την καλύτερη χρησιμοποίηση όλου του εναέριου χώρου. Καταλήγουμε λοιπόν σε μια προβληματική σε σχέση με μια συνεργασία μεταξύ των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών για τον ενάριο χώρο και ιδίως για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της αεροναυτιλίας όπως και στην περίπτωση της ε, έκθεσης Τάραν προηγουμένως νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει εδώ η ίδια λογική να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους στρατιωτικούς πόρους οι οποίοι είναι σημαντικοί για να μπορέσουν να βοηθήσουν και σε άλλους τομείς. Και επομένως η λογική αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί. Γιατί όλα αυτά ξεκινούν από το γεγονός ότι σε όλες τις χώρες μας ο στρατιωτικός τομέας έχει πάρα πολλά ε, στοιχεία, πάρα πολλού πόρου και εξοπλισμό που θα μπορούσε να είναι πρόσφορος για να χρησιμοποιηθεί και στον πολιτικό τομέα. Όπως είπα λοιπόν και στον κύριο Ταράν στο προηγούμενο θέμα, θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Να χρησιμοποιήσουμε τον στρατιωτικό τομέα για να προστατεύσει και την ασφάλεια στον πολιτικό εναέριο χώρο. Αυτή είναι λοιπόν μια λογική που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και από εμά, επειδή εμείς ασχολούμεθα τώρα με τον πολιτικό ε, εναέριο χώρο, να ενισχύσουμε την εποπτεία και την ασφάλεια σε αυτό το τομέα με, στρατιω... με τη χρήση στρατιωτικών πόρων και όχι να έχουμε περαιτέρω επενδύσεις μόνο και αποκλειστικά σε στρατιωτικά μέσα και στρατιωτικές ε, ε λειτουργίες για την προστασία του εναέριου χώρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Κρόνεμπερκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και θα πρέπει να πετύχουμε συνεργασία πολιτικού και σχετικού τομέα και στους ουρανούς. Ένα ερώτημα έχω για τον εισηγητή. Τι θα συμβαίνει με τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου καλύπτει και το θέμα ρωσικών αεροσκαφών που μπαίνουν σε φιλανδικό εναέριο χώρο. Ποιος παρακολουθεί, ποιος χειρίζεται αυτές τις δραστηριότητες. Αν υπάρχει αυτή η νομοθεσία για τον κοινό εναέριο χώρο. Παραβίαση λοιπόν εθνικού εναερίου χώρου. Αυτό με προβληματίζει. Και πώς θα αντιμετωπιστεί. Είναι κοινό πρόβλημα ή είναι εθνικό. Uh, Έχω και εγώ μια ερώτηση χτες συζητήσαμε τον Γαλιλαίο. Έναν άλλο τομέα για συνεργασία πολιτικού και στρατιωτικού τομέα, τεράστια ποσά απαιτούνται και εδώ έχουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και τα δύο είναι παλιά προγράμματα και τα δύο συνεπάγονται τεράστιο κόστος. Αυτή την περίοδο πιστεύω ότι είναι δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει ε, και τα δύο προγράμματα. Ακόμα και το 2007 συζητήθηκε το ΣΕΖΑΡ. Ε, υπάρχει σαφής προσέγγιση από πλευρά θετικής. Πώς θα χρησιμοποιηθεί ο ενίος ευρωπαϊκός ουρανός και πώς οι στατιωτικοί μπορούν να συνεργαστούν με τον πολιτικό τομέα. Η ερώτηση απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους και τους κοιόδης εισηγητές, τους συναδέλφους, για την συμβολή τους και την αξιολόγησή τους του σχεδίου εκθέσεως. Συμφωνώ ότι δεν έχουμε το κείμενο της καθήλυνα αρμοδίας επιτροπής. Δεν το έχω ούτε εγώ. Χρειάζεται ενδελεχέστερη ανάλυση το θέμα. Πρέπει να αλλάξουμε και τις προθεσμίες, ούτως ώστε να δούμε και ποια είναι η άποψη της καθήλυνα αρμοδίας επιτροπής. Δεν χρειάζεται περαιτέρω υπογράμμιση ε, ενό σημαντικού παράγοντα, του βασικού στοιχείου που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή της συνεργασίας του πολιτικού με το στρατιωτικό τομέα. Γιατί το λέω αυτό. Διότι δίνει μια ανάσα, δεύτερη ανάσα στο όλο πρόγραμμα. Ανοίγει, δημιουργεί δυνατότητες για αποτελεσματικότερη χρήση του ευρωπαϊκού εναερίου χώρου. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική όθηση στο πρόγραμμα. Πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα, το ταχύτερο δυνατόν, για να πετύχουμε τα ευκταία αποτελέσματα. Να τονίσω ότι χρειάζεται ωστόσο συντονισμός υπήρχε, είναι πολύ θετική συνέπεια, ε, έχει πολλές θετικέ συνέπειες η ιδέα εφαρμογή του ΕΕ, Χρειάζεται συνεργασία, συμφέρει το στρατιωτικό τομέα, χρειάζεται συνεργασία στο στρατιωτικού και πολιτικού τομέα. Σημαντικός είναι ο συμπληρωματικός εναέριος χώρος, ο πρόσθετος εναέριος χώρος και ευελιξία χρήσεως του εναερίου χώρου. Στις συναντήσεις εργασίας που είχα με συναδέλφους έντα, εγώ τόνιζα πώς απογοητευμένος ήμουνα σαν πολίτης που έβλεπε ότι καμιά φορά έκλεινε ο εναέριος χώρος ή κάποια κομμάτι του εναέριου χώρου λόγω θετικών ασκήσεων. δεν υπήρχε τεχνολογικός τρόπος για τον σωστό συνδυασμένο ε, τρόπο για συνδυασμένη χρήση του εναερίου χώρου. Χρειάζεται αυτή η συνεργασία. Χρειάζεται συνεργασία για να είναι αποτελεσματική όπως ήταν μέχρι τώρα, αλλά να είναι πιο παραγωγική στο μέλλον. Οπότε είναι ευπρόσδεκτες οι πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι σχετικέ. Για τις παραβιάσεις εναερίου χώρου δεν νομίζω ότι είναι το βασικό μας θέμα, διότι το έθεσε η Φιλανδή συνάδελφος. Παραβίαση εναερίου χώρου όσον αφορά τους στρατιωτικούς είναι κάτι διαφορετικό. Θέλω να ακούσω ποια είναι η άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που έχω να πω σε αυτό το στάδιο είναι αυτό που τόνισαν και συνάδελφοι. χρειάζεται να βρούμε τρόπους για να βοηθήσουμε τους αιτητικούς. Αυτό πάντα τονίσουμε. Δεν θα είναι εύκολο το εγχείρημα, διότι πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες διαφόρων χωρών. Με διαφορετικά αεροσκάφη, διαφορετικό εξοπλισμό, και ταυτόχρονα μας ενδιαφέρει όλους αυτή η συνεργασία. Όπως προανέφερα δεν προβλέπονται σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά ε, το πολιτικό, τις πολιτικές αερομεταφορές. Χρειάζεται όμως κάποια ενίσχυση από πλευράς του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μπορούν να βοηθηθούν χώρες που θα αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, γιατί περνάμε και χαλεπούς καιρούς. Και θα δοθούν και κίνητα ταυτόχρονα σε χώρες για να εφαρμόσουν ταχύτερα το πρόγραμμα αυτό. Για να πετύχουμε αποτελέσματα, να έχουμε πραγματικό ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ρώση, εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να απαντήσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει έχω να απαντήσω. Η πρώτη είναι μια τεχνική φύσεως ερώτηση για την πιθανή παραβίαση αέριου χώρου. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ διαχείρισης της κίνησης και της άμυνας. Είναι δύο διαφορετικά στοιχεία. Το πρώτο αφορά τον ενίο ευρωπαϊκό ουρανό και τον τεχνολογικό πυλώνα, το ΣΕΖΑΡ, αλλά υπάρχει μια σχέση με την άμυνα σε κάποιο βαθμό, διότι όταν ε, ζητάμε από το στρατιωτικό τομέα να κάνει μια ε, διείσδυση, αυτό θα ε, επηρεάσει και το δίκτυο των μεταφορών και φυσικά αυτό πρέπει να το δούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν έχει αλλάξει τίποτα για το ποιος έχει την ευθύνη. Η ευθύνη για τον εναέριο χώρο είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και έχουν εμπιστευτεί ε, το στρατιωτικό σκέλος στο ΝΑΤΟ. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό ρυθμίζεται και από το άρθρο 28 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Όλα είναι σαφή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία λοιπόν από αυτού και δεν υπάρχει καμία ανάγκη ε, να ε, συζητήσουμε τίποτα περαιτέρω για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα το κόστος ε, για το ΣΕΖΑΡ, εδώ πρέπει να είμαι σαφής. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να επεκταθώ λίγο περαιτέρω στο ΣΕΖΑΡ και στο τι αφορά. δημιουργήθηκε για μια διαδικασία ορισμού, ανάπτυξης και από εκεί και πέρα ε, επιπλέον εξέλιξης. Η διαδικασία αυτή η τελευταία θα στοιχήσει περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό φυσικά είναι το αρνητικό σκέλος. και θα πρέπει να εφαρμοστεί βάση των πραγματικών αναγκών ε, του ε, Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειων Μεταφορών. Δηλαδή δεν θα εφαρμοστεί τεχνολογία απλώς και μόνο για να χρησιμοποιήσουμε τη νέα διαθέσιμη τεχνολογία. Θα εφαρμόσουμε αυτό που χρειάζεται διότι πραγματικά έχει αυξηθεί η κίνηση στους ουρανούς. Το βασικό τώρα ε, σχέδιο του ΣΕΖΑΡ λαμβάνει υπόψη και τις πολιτικές αλλά και τις στρατιωτικές ανάγκες. Και όπως σας είπα την περασμένη ε, Παρασκευή, ο αρχηγός Αμυνάς ε, συναντήθηκε με τους αρμοδίους και πλέον υπάρχει συνεννόηση, προσπαθούν να συνεργαστούν με τους πολιτικούς τους εταίρους, ώστε να υπάρχει έγκαιρη και συγχρονισμένη εφαρμογή του ΣΕΖΑΡ, διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν δεν εφαρμοστούν οι τεχνολογίες αυτές με συγχρονισμένο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όλα αυτά θα είναι εις βάρος φυσικά και της απόδοσης αλλά και της αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος. Γι' αυτό λοιπόν και το στρατιωτικό σκέλος θα πρέπει να συμμετέχει στο σχεδιασμό της ανάπτυξης ε, ε, και της εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας. Ελπίζω να σας απάντησα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι κάπως ε, παράδοξο να συζητάμε μια γνωμοδότηση χωρίς να είναι διαθέσιμη η επί έκθεση. Ξέρουμε ότι θα καθυστερήσει λιγάκι η έκθεση του κυρίου Φώστα γιατί έχουν προβλήματα με τη μετάφραση, αλλά η προθεσμία της τροπολογίας είναι 16 Μαΐου το μεσημέρι. 29 Μαΐου θα εξετάσουμε και πάλι την γνωμοδότηση και η ελπίδα μας είναι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη ημερομηνία, στις 7 ή στις 18 Ιουνίου θα εγκριθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και μετά στις 9 ή 10 Ιουλίου στην Επιτροπή Μεταφορών και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Και σας υπενθυμίζω στις 8 Μαΐου ότι θα έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση το πρωί και η επόμενη τακτική μας συνεδρίαση είναι 29 Μαΐου πρωί αλλά και απόγευμα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο στην ημερήσια διάταξή μας. Κλείνω λοιπόν την συνεδρίαση ευχόμενη σε εμά μια πολύ καλή ξεκούραση το Σαββατοκύριακο.